Προχωράμε λοιπόν στις επεξηγήσεις ψήφου ζητώντας στις συναδέλφους και τους συναδέλφους να ε, εγκαταλείψουν την αίθουσα χωρίς πολύ θόρυβο και χωρίς πολλές συζητήσεις. Η κυρία Σβίρμπουρν για ένα λεπτό. Η αλληλεία, παρά το ότι έχει μειωθεί, αλλά έχει μεγάλη σημασία για τους ψηφοφόρους στην Ουαλία, συμβάλλει στην ευρύτερη οικονομία. Χαιρετίζω την έκθεση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας. Είναι ένα από τα μέσα που θα βοηθήσει την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινή αλληλευτική πολιτική, δηλαδή να υπάρξει αηφορία των ε, ηχθειών με αυτά τα επιπλέον ε, χρήματα η έκθεση προτείνει το Ταμείο να δώσει χρήματα στην οικονομία για να συνεχιστούν τα προγράμματα. Η Αλία επίσης βοηθάει και τον τουρισμό, ιδιαίτερα στη Δυτική Ουαλία που λαμβάνει χρήματα από το Ταμείο Συνοχής. Πρέπει λοιπόν το Ταμείο αυτό να βοηθήσει τις περιοχές που το, χρειάζονται περισσότερο, τους ε, αλληλείς να ενισχύσει και τον τουρισμό και τη διαφοροποίηση της οικονομίας. Ευχαριστώ. Για τις υπό... επόμενες παρεμβάσεις παρακαλώ τους συναδέλφους να μιλούν με αργότερο ρυθμό γιατί διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν μεγάλες δυσκολίες ε, οι διερμηνείς. Το λόγο έχει η κυρία Άννα Ρόσμπαχ. formand det er grundlæggende marked. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει μια αντίφαση με την εσωτερική αγορά. Η προσπάθεια ενίσχυσης ενός συγκεκριμένου τομέα της ελίας ε, τον φέρνει ως τομέα εξαρτημένο, κάτι που στρεβλώνει την ενή αγορά. Πάντως η τελευταία πρόταση είναι βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες. Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη και την περιβαλλοντική διάσταση. Είναι σημαντική η ύπαρξη ενός τέτοιου ταμείου, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας, αλλά θα πρέπει οι πιστώσεις του ταμείου αυτού να συμβάλλουν στην ενίσχυση της ε, ε, οικονομικής δραστηριότητας. Ευελπιστώ ότι στο μέλλον θα καταργήσουμε επιδοτήσει που έχουν αρνητικό χαρακτήρα στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ είμαι υπέρ μια ελεύθερη ενιαία αγορά. Αυτή είναι η βέλτιστη λύση και για του καταναλωτέ, αλλά και για του φορολογούμενου. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Ήβα Τζανίκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε σε ένα πλαίσιο γενικευμένης οικονομικής κρίσης που βεβαίως δημιουργεί ιδιαίτερο πρόβλημα και στις παράκτιες κοινότητες της Ευρώπης νομίζω ότι είναι η στιγμή για να χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας. Πολύ συχνά τα χρήματα τα οποία δόθηκαν πολύ συχνά αφορούσαν την καταστροφή σκαφών. Ε, θα ήθελα αυτή τη στιγμή να ζητήσω να ε, εντείνουμε τις προσπάθειές μας έτσι ώστε να διατηρηθεί η οικονομική δραστηριότητα της Αλίας και επίσης ε, να διευκολύνουμε την πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Εγώ έδωσα τη θετική μου ψήφο στην έκθεση της κυρίας Φερέιρα ε, με την ελπίδα ότι μέσω της ψήφου αυτή θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη βοήθεια που δίνεται στα κράτη και στις παράκτιες κοινότητες έτσι ώστε να συνεχιστεί η αλληλευτική δραστηριότητα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τζανίκη. Η κυρία Αντζελίλη. Κυρία Αντζελίλη, παρακαλώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε το είπαν και άλλοι πριν από μένα, το σενάριο γενικευμένης ε, κρίσης ε, το, το οποίο έρχεται μετά από χρόνια σημαντικής παρακμής ε, και δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας μεταξύ των οποίων και η αλληλεία για την Ιταλία αλλά και για άλλες χώρες όπως η Ελλάδα α πούμε η αλληλεία αποτελεί αφενός ένα εισόδημα αφετέρου ε, σημαντικό οικονομικό παράγοντα για την οικονομική ζωή πολλών περιοχών. Ε, εγώ θέλησα να στηρίξω την πρόταση της Επιτροπής έτσι ώστε να δοθούν επιπλέον 10% ποσοστά συγχρηματοδότησης ε, όσον αφορά τα καταπροτεραιότητα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλίας έστω ε, πρόσκαιρα έτσι ώστε να δημιουργήσουν κάποιο κίνητρο σε ιδιωτικούς ε, και δημόσιους επενδυτές έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν σωστά τα κονδύλια τα οποία θέτει στη διάθεσή του η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Αντζελίλη. Πυρίλο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε ψήφισα υπέρ της εκθέσεως ε, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας θεωρώντας ότι είναι απαραίτητη έτσι ώστε να ε, διευρυνθούν τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλίας και ε, που απευθύνονται σε όλες τις χώρες. Συμφωνώ λοιπόν και συμφώνησα και με την πρώτη ανάγνωση. Πολύ καλά έκανε η Επίτροπος κυρία Δαμανάκη η οποία με επίγουσα διαδικασία προχώρησε στην την προσπάθεια ε, να ξεπεραστούν τα προβλήματα της ελευτικής ε, διαδικασίας ε, που έχει φτάσει σε ιστορικά χαμηλά. Θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιηθούν σωστά τα χρήματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλείας, χρησιμοποιώντας και αυτό το περιθώριο του επιπλέον 10% όσον αφορά τη συγχρηματοδότηση, έτσι ώστε ε, να μπορέσουμε ε, σε αυτήν την εκστρατεία να χρησιμοποιήσουμε, σε αυτή την προγραμματική περίοδο, να χρησιμοποιήσουμε και χρήματα τα οποία έχουν περισσέψει από την προηγούμενη περίοδο. Και αυτό για το καλό της αλλιευτικής δραστηριότητας και της αλλίας γενικότερα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πυρίλο. Πίτερ Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ με πάλι χαρά ενέκνα αυτό το ψήφισμα. Είναι η σωστή απάντηση στα τωρινά προβλήματα που έχουμε στα κράτη-μέλη. Όλοι προσπαθούμε να βοηθήσουμε την οικονομική συγκυρία. Δύο προβλήματα υπάρχουν. Το ένα είναι ότι οι χώρες δεν έχουν επαρκείς πιστώσεις. Το άλλο είναι ότι δεν λειτουργεί η προχρηματοδότηση πολλών προγραμμάτων. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Η προχρηματοδότηση να βελτιωθεί, στην αρχική φάση δηλαδή, και πρέπει φυσικά να υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να είναι παράδειγμα και για άλλα ταμεία, αυτό το Ταμείο Αλίας. Παρακαλώ λοιπόν τα αποτελέσματα να δούμε αν μπορούμε να τα εφαρμόσουμε και σε άλλα προγράμματα και ταμεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριο Τάνοκ. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ ψήφισα μαζί με την ομάδα μου υπέρ της έκτης Φεραίρα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας. Τα προγράμματα όπως το EFF, δηλαδή το Ταμείο Αλίας, είναι πολύ χρήσιμο στα κράτη-μέλη που έχουν υποφέρει περισσότερο από την κρίση. Είναι πολύ δύσκολο γιατί είναι δύσκολο να υπάρξει συγχρηματοδότηση προβλέπεται πρόταση επιτροπή που θα επιτρέψει να ενισχυθούν οι πληρωμέ προ τι χώρε που έχουν αντιμετωπίσει τι περισσότερε δυσχέρειε από την οικονομική χρήση. Δηλαδή αυτέ τι χώρε που ήδη λαμβάνουν και άλλη στήριξη. Χαιρετίζουμε το ότι το ποσό που θα συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι περισσότερο από την αρχική πρόταση της Επιτροπής, δηλαδή πάγωμα του προπολογισμού όπως είχαμε ακριβώς ζητήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Τάνοκ. Το λόγο έχει ο κύριος Νίκολσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ υπερψήφισα την έκθεση Φεραίρα. Στην παρούσα χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση που μαστίζει την Ευρωζώνη θα πρέπει να χαράξουμε το δρόμο για μια ομαλή εφαρμογή των διαρθρωτικών προγραμμάτων όπως αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Υπερψηφίζοντας την έκθεση αυτή βοηθούμε την μεταφορά κονδυλίων στις τοπικές ε, κοινότητες και στις τοπικές οικονομίες. Είμαι υπέρ και των μηχανισμών που θεσπίζονται και που ε, προβλέπουν ε, ενισχυμένες πληρωμές προς χώρες που έχουν χρηματοοικονομικές δυσκολίες εφαρμογής των προγραμμάτων, όπως είναι η Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία και στη Βόρεια Ιρλανδία. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν τι παρενέργειε αυτή τη οικονομική ε, ύφεση και νομίζω ότι αυτό είναι και στόχο ε, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλία. Ελπίζω να είναι θετικά τα αποτελέσματα. Άλλωστε, δεν υπερβαίνουμε πάνω από 10% τα ανώτατα όρια που προβλέπονται από τον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλία. Σα ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριο Καμίνσκι. Κύριε Πρόεδρε, θα ε, ήθελα να πω ότι υπερψήφισα ε, θερμά υπέρ ε, της έκθεσης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο γιατί κρίνω ότι η Αλία είναι σημαντικός οικονομικός κλάδος της ευρωπαϊκής οικονομίας. Και η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει την ελαστικότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέναντι στην κρίση που μαστίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί Απ' τη μια δεν λαμβάνουμε υπόψη τις προσδοκίες ε, των ε, φορολογουμένων, αλλά μερικές φορές ε, δείχνουμε κάποιο ορθολογισμό στις, και ρεαλισμό στις αποφάσεις μας. Οι αποφάσεις αυτές δεν έχουν μόνο οικονομική διάσταση, αλλά και υγειονομική διάσταση. Μιλήσαμε και για την για την επιδημία του διαβήτη. Η, διατροφή με ψάρια είναι πολύ σημαντικός παράγοντας υγιεινής διατροφής και νομίζω ότι έτσι θα βελτιώσουμε και την υγεία των συμπολιτών μας. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Κέλλη για ένα λεπτό. Mr. Kelly. Sorry, President, I Κύριε Πρόεδρε, δεν ζήτησα το λόγο για επεξήγηση ψήφου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο εγώ ψήφισα υπέρ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ελίας, υπέρ της έκθεσης Φερέιρα. Συγγνώμη κύριε Κέλλη. Απλώς είδα το όνομά σας στον κατάλογο με τις επεξηγήσεις ψήφου. Καλώς, περνάμε στις επεξηγήσεις ε, ψήφου για την έκθεση Quisthout Revol. Το λόγο έχει η κυρία Σουίνμπερν. E Ευχαριστώ. Εφόσον απογορεύσαμε τις εισαγωγές από βοήων προϊόντων με, από τις Ηνωμένε Πολιτείες και τον Καναδά είχαμε την έγκριση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για κυρώσεις κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πολλές επιπτώσεις. Χαίρομαι λοιπόν που υπάρξει ένα, ε, μια επίλυση του προβλήματος αυτού. Είναι σημαντικό το ότι έχουμε τώρα μια αυτόνομη ε, ποσόστοση για υψηλού επίπεδου εισαγωγές βοηδών θα μας επιτρέψει αυτό να ξαναχτίσουμε τις εμπορικές μας σχέσεις στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ κυρία Βίρμπουρ. Ο κύριος Άνναν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πριν από 40 χρόνια το Ηνωμένο Βασίλειο ψήφισε να μπει στην κοινή αγορά. Δεν νομίζω ότι καταλάβαμε ούτε τότε ούτε τώρα την διαφορά μεταξύ μιας ελεύθερης αγοράς και μιας τελωνιακής ένωσης. Μια ελεύθερη αγορά εμπορίου σημαίνει ότι τα αγαθά, το κεφάλαιο υπηρεσίες μπορούν να κυκλοφορήσουν χωρίς ε, περιορισμούς. Τέτοια σχέση έχουν οι Ελβετοί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα πάνε πολύ καλά. Σε μια τηλεοναϊκή ένωση βεβαίως σύρεται κανείς σε μια κοινή εμπορική πολιτική και κοινά, κοινό εξωτερικό δασμολόγιο. Αυτό έχει ολέθρες επιπτώσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο που το μεγαλύτερο τμήμα του εμπορίου του το κάνει προς μη ευρωπαϊκές αγορές. Είμαστε σε μια αγορά παρόμοιων εκβιομηχανισμένων οικονομιών και έχουμε αποκοπεί από τους παραγωγούς πρώτων υλών. Έχουμε περιοριστεί, και το επαναλαμβάνω, σε μια ε, ιδιαίτερα πολυπληθή και φθήνουσα ε, Ευρωπαϊκή Δασμολογική Ένωση. Πραγματικά οι προηγούμενοι μας έλαβαν μια πολύ λανθασμένη απόφαση. Ευχαριστώ κύριε Άννα. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Ήβα Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θετικά ψήφισα για την έκθεση αυτή που έχει στόχο την ευθυγράμμιση κάποιων νομοθετικών πράξεων ε, της εμπορικής εξωτερικής πολιτικής ε, με την επιτροπολογία καθώς επίσης και κάποιες νομοθετικές πράξεις όσον αφορά ε, την γεωργική πολιτική. Είναι σωστές οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε μια στιγμή ιδιαίτερης κρίσης όπου το Made in Italy ας πούμε θα πρέπει να μας δώσει περισσότερες ευκαιρίες πιστεύουμε ότι τέτοιου είδους πρακτικές μπορούν να να βοηθήσουν τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Ε, οι εμπορικές ε, πρακτικές ε, στρέβλους του ανταγωνισμού από εξωτερικούς μη ευρωπαίους ανταγωνιστές μπορεί να δυναμητήσουν την προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Τάνοκ. Κύριε Πρόεδρε, με τις δυσχέρειες που υπάρχουν στο διατλαντικό εμπόριο ζωικών προϊόντων είχαμε αυτή τη διαμάχη για το χλώριο στα πουλερικά και το πρόβλημα με τις ορμόνες. Πιστεύουμε ότι αυτός ο κανονισμός θα ενισχύσει τους ζωτικούς δεσμούς εμπορίου, τους διατλαντικούς και θα βελτιώσει πρόσβαση στην αγορά και στις δύο πλευρές, οπότε θα έχουμε περισσότερη εμπιστοσύνη. Τα προϊόντα που είχαν ε, επηρεαστεί από την απαγόρευση για τις ορμόνες ήταν λίγα. Είχαμε επιπτώσεις από τις αντιδράσεις των ΗΠΑ. Ελπίζουμε αυτές οι κυρώσεις των ΗΠΑ να αρθούν και να καταργηθούν οι φραγμοί η πρόταση που προτείνεται για κανονισμό θα βοηθήσει τις ε, μακροχρόνιες διατλαντικές εμπορικές σχέσεις με οικονομικά ωφέλη και στις δύο πλευρές. Οι πολιτικές και εμπορικές μας σχέσεις με τις ΗΠΑ πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητά μας λόγω των κοινών δημοκρατικών αξιών μας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος Νίκολσον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπερψήφισα, υπερψήφισα το θέμα αυτό, αν και είχα κάποιες ανησυχίες αρχικά γιατί μακροπρόθεσμα πιστεύω ότι η έκθεση αυτή θα δημιουργήσει μια κατάσταση όπου θα κερδίσουν και οι Ηνωμένε και ο Καναδά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση δημιουργεί τρόπο να ξεπεράσουμε την καταστροφική δυναμική των ε, εμπορικών κυρώσεων και των δασμών που ξεκίνησαν στη δεκαετία του 80 λόγω της απαγόρευσης ε, βοήων και βοηών προϊόντων επειδή είχαν ορμόνες. Αυτοί οι δασμοί είχαν επιπτώσεις πάνω από 116 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Οι ΗΠΑ και ο Καναδάς πρόσφατα ήραν τις κυρώσεις τους για να δημιουργήσουν μια ποσόστοση για υψηλής ποιότητας, ποιότητας ε, βοηδών προϊόντων που θα μπορούν να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει αυτό το μέτρο. Η έκθεση αυτή θα δώσει 20.000 το χρόνο βοηδή προϊόντα υψηλού επίπεδου η επίλυση αυτής της ε, διαφωνίας για τις ορμόνες θα εμβαθύνει την οικονομική και πολιτική ενοποίηση μεταξύ αυτών των δύο περιοχών. Ευχαριστώ κύριε Σκαμίνσκι. Κύριε Πρόεδρε, η διαμάχη ε, που μέχρι στιγμής ισχύει ελπίζω σήμερα να ολοκληρωθεί. Ξεκίνησε το 1998. Τότε η εξαγωγής έχασαν ε, πάνω από 116 εκατομμύρια ε, δολάρια το χρόνο εξαιτία τη απαγόρευση ε, εξαγών από την Ευρωπαϊκή Ένωση προ ε, τι Ηνωμένε Πολιτείε. Ήταν τα αντίπεινα των Ηνωμένων Πολιτειών για τι απαγορεύσει που εφάρμοζε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ είμαι υπέρμαχο τη ε, ελεύθερη αγορά και πιστεύω ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε θα πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στι φυτογενομικέ διατάξει που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και εμεί θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στι διαδικασίε ασφάλεια των τροφίμων που ισχύουν στι Ηνωμένε Πολιτείε. Φαίνεται ότι σήμερα ε, πραγματοποίησαμε ένα πολύ καλό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και ευελπιστώ ότι η ΕΠΑ θα δώσουν μια θετική απάντηση στην ε, χειρονομία καλής θέλησης των Ηνωμένων, των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ κύριε Καμίνσκι. Περνάμε στην επόμενη έκθεση της κυρίας Κβίστ Χαουτ. Το λόγο έχει η κυρία Σουίνμπερν. Πρόκειται για τεχνική έκθεση. Ενημερώνει τι διαδικασίε για να λάβουν υπόψη το νέο γιατί μετά την ένταξη, μετά την αρχή ισχύω της συνθήκη της Λισαβόνας Αλλά θα έχει επιπτώσεις στους κανονισμούς και το περιεχόμενό του. Ο ρόλος που έχει το Κοινοβούλιο σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε το ρόλο μας αυτό πολύ σοβαρά. Στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή περάσαμε πολύ χρόνο συζητώντας εάν κάτι είναι καθαρά τεχνικό και πρέπει να είναι εφαρμοστικό μέτρο ή αν θα πρέπει να είναι μια συγκεκριμένη πράξη την οποία μπορούμε κατόπιν να ανακαλέσουμε. Στα θέματα τη εμπορική πολιτική είμαι σίγουρη πω η ισορροπία είναι πολύ δύσκολη όπω είναι και σε θέματα οικονομικών αγορών. Θετικά πιστεύω ότι η έκθεση όπω είναι έχει επιτύχει τη σωστή ισορροπία. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Μουσκαρδίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κανονισμός κατά του Ντάμπικ ε, αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη προσπάθεια εξορθολογισμού. Ε, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι η κοινή εμπορική πολιτική για να είναι αποτελεσματική και να μην ε, είναι επιβλαβής για τους παραγωγικούς τομείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να σέβεται τους κανόνες και μάλιστα οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να ισχύουν για όλους τους συνομιλητές. Το ζήτημα, ο κανόνας της διόρθωσης των τιμών είναι πολύ σημαντικές. Θα πρέπει να δείξουμε ενεργητικότητα και αποτελεσματικότητα. Γι' αυτό λοιπόν ε, εμείς θέλουμε να ε, υπάρξει πλήρης κάλυψη όλων αυτών των διαδικασιών ε, αντι-dumping που δεν πρέπει να ξεπερνούν τους 15 μήνες. Δεν θέλουμε να αποδυναμώσουμε όπως λέει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα όσα προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας και τα οποία είναι απαραίτητα έτσι ώστε να διασφαλίσουν τους κανόνες, να διασφαλίσουν τα συμφέροντα των τελικών καταναλωτών καθώς επίσης ε, ε, και την μη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Μουσκαρντίνη. Δεν βλέπω να είναι εδώ η κυρία Τζανίκη και επομένως περνάμε στον επόμενο ομιλητή. Σου, σούστα, λείπει. Και επομένως φτάνουμε στον κύριο Καμίνσκι. Κύριε Πρόεδρε, με μεγάλη υπευθυνότητα ψήφισα μαζί με την ε, πολιτική μου ομάδα υπέρ της έκθεσης Κβίστκαου Ροβόλ. Προβλέπει κάποιες τεχνικές διατάξεις ε, που συνδέονται και με το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σταδιακά εφαρμόζει αυτές τις ε, συστάσεις και προσαρμόζεται στη, στον ενισχυμένο του ρόλο μετά την συνθήκη της Λισαβόνας. Φυσικά εγώ ε, είμαι αναφεδόν υπέρ ε, της διαδικασίας αυτής και χαίρομαι ότι ε, χαίρομαι που μόνο με ε, ενισχυμένη πλειοψηφία μπορούν να, προ, να αναχαιτιστούν κάποιες προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. είχαμε την πρόσφατη περίπτωση των μέτρων αντιντάμπικ. Θέλουμε κάποιους μηχανισμούς για να προασπίσουμε την εσωτερική αγορά, την ευρωπαϊκή αγορά και να διαφυλάξουμε και τους πολίτες μας. Ευχαριστώ κύριε Καμίνσκι. Το λόγο ο κύριος Μπιέλαν. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, παρά κάποιες επιφυλάξεις και φόβους που είχα για τις ατελείς διαπραγματεύσεις με τα κράτη-μέλη, αποφάσισα τελικά να ψηφίσω υπέρ της έκθεσης. Ο κανονισμός αυτός προβλέπει την προσαρμογή κάποιων διατάξεων για την κοινή, την κοινή εμπορική πολιτική στι ε, διατάξει τη συνθήκη Λισαβόνα. Για παράδειγμα, κάποιε εκτελεστικέ διατάξει που αφορά την ομοιόμορφη μεταφορά του κοινοτικού δικαίου σε όλε τι εθνικέ νομοθεσίε, αντικαθιστώντα την ισχύουσα διαδικασία τη επιτροπολογία. Πολύ σημαντικό μηχανισμό εδώ θα είναι κάποιε διαδικασίε συμβουλευτικέ και ελεκτικέ. Η εφαρμογή των κατεξουσιοδότηση πράξεων επιτρέπει κατάλληλο έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στον τομέα αυτό. Πολύ καλή πρόγνωση, ε, ε, ε, πολύ καλό ιονό είναι η λήψη υπόψη των συστάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα τη μείωση ή την κατάργηση δασμών σε προϊόντα κάποιων δασμολογικών θέσεων της κοινής του ενιαίου δασμού. Ελπίζω ότι με τη διαδικασία αυτή θα ενισχυθούν οι εμπορικέ ε, ανταλλαγέ μεταξύ των χωρών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και με, χώρες, με τρίτε χώρε προ όφελο και των συμπολιτών μα. Περνάμε στην έκθεση Λαβία και δίνω το λόγο στην κυρία Σουίνμπερν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπω και η πολιτική μου ομάδα, του Ευρωπαίου Συντηρητικού και Μεταρρυθμιστέ, θα θέλω να μειωθεί αρκετά ο προπολογισμό. Δεν μπορώ να υποστηρίξω αυτή την έκθεση, γιατί υποστηρίζει έναν ακόμη μεγαλύτερο κοινοτικό προπολισμό που δεν μπορώ να αιτιολογήσω αυτή τη στιγμή στους ψηφοφόρους μου στην Ουαλία. Πολλά κράτη-μέλη εφαρμόζουν σκληρά μέτρα λιτότητας που είχαν καταστροφικές επιπτώσεις στην ε, ζωή και το εισόδημα των ατόμων. Θα ήταν εντελώς αδικαιολόγητο να υποστηρίξουμε οποιαδήποτε αύξηση στον προπολογισμό της Ένωσης. Όλοι οι θεσμοί πρέπει να επιδείξουν την δυνατότητα να μειώσουν του προπολογισμού τους λόγω, λόγω της κρίσης. Ο προπολογισμό του 2013 θα πρέπει να μην έχει καμία αύξηση. Ευχαριστώ. Χάναν. Τρία είναι σίγουρα πράγματα στη ζωή. Ο θάνατος, η φορολογία και η συνεχής αύξηση του προβλημού της Ένωση. Αυξάνεται συνέχεια η συμβολή των κρατών μελών, όλα τα 27 κράτη-μέλη, ενώ προσπαθούν να μειώσουν την τους, την, ε, τον εθνικό τους προπολογισμό ακυρώνουν αυτή την προσπάθεια μέσω υψηλότερη συμμετοχή ε, στον κοινοτικό προπολογισμό μα. Λένε ότι τα χρήματα αυτά δημιουργούν θέσει εργασία, ενθαρρύνουν την ευημερία. Όσοι δεν ξέρουν αγγλικά μπορούν να δουν το άρθρο του Φρέντρικ Μπάστια για το κόστος που υπάρχει και το αόρατο. Κάθε ε, χρήμα που παίρνουμε για να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να ε, δημιουργηθεί πραγματικός ε, πλούτος. Όλοι αυτοί οι γραφειοκράτες, όλοι αυτοί οι ρυθμιστικοί μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ουσία τι αποδεικνύουν. Πώ μπορούμε να συνεχίσουμε με ένα τέτοιο σύστημα όπου για να πληρώσουμε για αυτόν τον συνεχώ αυξανόμενο κοινοτικό προπολογισμό, όσο μιλάω, οι ψηφοφόροι μου έδωσαν στην Ένωση περίπου 120 λίρε. Οπότε σταματάω να μιλάω και κάθομαι. Ευχαριστώ κύριε Χάναν. Ο κύριος Αντωνιώτση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πριν από την επεξήγηση ψήφου θέλω να σας πω ότι φοράω αυτό το μπλουζάκι για να ζητήσω την έγκριτη παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελεύθερηση του Μασιμιλιάνο Λατόρες και του Σαλβετόρο Τζιρόνε, τους δύο στρατιωτικούς ε, Ιταλούς που κρατούνται από τους πειρατές. Ε, σχετικά με, τον, με τις Γενικές Κατευθυντήριες Γραμμές και τον Προϋπολογισμό 2013 είναι αυτές οι οποίες θα καθορίσουν ε, και την, τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, στην λόγω έκθεση καθορίζονται τα σημεία κλειδιά για την αναδιάρθρωση της ευρωπαϊκής οικονομίας έτσι ώστε να μπορέσει να ξεφύγει από την στασιμότητα που προκαλεί αυτή η διαρκής οικονομική κρίση. Υπάρχουν νέα εργαλεία τα οποία βοηθούν ακολουθούν τα κράτη-μέλη ε, αλλά και ε, ενέχεται και η ε, υπόσχεση ότι θα μπορέσουν να βρεθούν λύσεις ξεπεράσματος της κρίσης που πλήττει αυτή τη στιγμή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ με την έκθεση του κυρίου Τζοβάνι Λαβία, κυρίως δε με το αίτημά του προς το Συμβούλιο να μην υπάρξουν τεχνητές περικοπές οι οποίες δεν θα λαμβάνουν υπόψη την δυνατότητα απορρόφησης, εγγενούς απορρόφησης των κονδυλίων και που θα επιβραδύνουν την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε ε, Αντωνιώτσι. Ε, βεβαίως συμμεριζόμαστε την έκκλησή σας ε, και εγώ προσωπικά και φαντάζομαι και πολλοί συνάδελφοι του συναδέλφου και ευελπιστούμε ότι από τη στιγμή που θα έχουμε σήμερα την ύπατη εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας θα μας δώσει και κάποιες πληροφορίες για αυτή τη δύσκολη και δραματική κατάσταση. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Μαρίνα Γιανακουδάκη. Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση αυτή ζητά συλλογικέ προσπάθειε για την ενίσχυση τη ευρωπαϊκή οικονομία. Στην πράξη σημαίνει περισσότερη Ευρώπη και περισσότερα χρήματα. Εγώ είμαι υπέρ τη ανάπτυξη και των θέσεων απασχόληση, αλλά δεν νομίζω ότι ο κατάλληλο τρόπο για να το επιτύχουμε κάτι τέτοιο είναι με περισσότερη Ευρώπη. Χρειαζόμαστε λιγότερη γραφειοκρατία, λιγότερου κανονισμού για να μπορέσουν να ευδοκιμήσουν οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει. Δυστυχώ χάσαμε μια ευκαιρία να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα. Θα έπρεπε να είχαμε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει περισσότερε επιδόσει με λιγότερα κονδύλια ανταποκρινόμενοι στην έκκληση των συμπολιτών μα για ένα πάγωμα του ευρωπαϊκού ε, προϋπολογισμό. Αλλά όπως συνήθως φοβηθήκαμε, γι' αυτό δεν μπορώ να υποστηρίξω την έκθεση. Ευχαριστώ κυρία Γιάννα Κουδάκη. Το λόγο κυρία Ντότς. Ευχαριστώ. Εγώ ψήφισα κατά της έκθεσης γιατί για μία ακόμη φορά η περαιτέρω οικονομική ολοκλήρωση θεωρείται ως προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ πιστεύω ότι αντί να είναι ο ακρογωνιός λίθος οποιοδήποτε ανάκαμψης ε, ε, η ολοκλήρωση ουσιαστικά είναι αυτό που υπονομεύει ε, την ευρωπαϊκή οικονομία και ενισχύει την καταβαράθρωση. Φαίνεται ότι εθελοτυφλούμε μπροστά στην πραγματικότητα. Δεν πρόκειται δυστυχώς η ανάκαμψη που επιζητούμε να λάβει χώρα με ικανοποιητικό ρυθμό. Η λιτότητα που έχει επιβληθεί σε πολλέ χώρε μέλη δεν θα πρέπει να. Ε, γιατί δεν πρέπει να έχει ένα αντίκτυπο και στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Τι αλαζονία δείχνουμε. Γιατί εμεί απαιτούμε περισσότερα κονδύλια από τα κράτη-μέλη προ την Ευρωπαϊκή Ένωση, προ τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Κάντε ό,τι λέω και όχι ό,τι κάνω. Αυτό φαίνεται ότι είναι το μήνυμα που δίνει πολύ συχνά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήρθε η ώρα να περιορίσουμε τις, ε, τις πατάλες του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, να προωθήσουμε την ανάπτυξη της, και την απασχόληση, αλλά πρώτα απ' όλα να δώσουμε εμείς το καλό παράδειγμα. Ευχαριστώ κυρία Ντότς. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ. Υπερψήφισα την έκθεση γιατί νομίζω ότι ο συγητής Τζοβάν Λαβία έκανε μια θαυμάσια εργασία, επέτυχε τους αναγκαίους συμβιβασμούς και γιατί νομίζω ότι όταν μιλάμε για στρατηγικούς στόχους, για μείωση της γραφειοκρατίας, άρα απευθυνόμαστε στην Επιτροπή, τη ζητάμε να χρησιμοποιήσει λιγότερα χρήματα. Είναι στρατηγικός στόχος, δεν μπορεί να επιτευχθεί από τη μια μέρα στην άλλη. Πρέπει να ξεκινήσουμε να το αντιμετωπίζουμε, να δούμε πώς οι κανονισμοί μας θα χρειάζονται λιγότερη γραφειοκρατία και θα προκαλούν, θα προκαλούν λιγότερη ανάγκη ελέγχου. Όμως θα ήθελα η τροπολογία Άλντε να εγκριθεί, δηλαδή ο προϋπολογισμός 2013 να ασχοληθεί περισσότερο με την ανάκαμψη μετά την αντιμετώπιση της κρίσης. Αυτό είναι έλλειψη, αλλά παρόλα αυτά την υπερψήφισα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τάκουλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, υπερψήφισα την έκθεση αυτή γιατί συμπεριλαμβάνει πολλά θετικά στοιχεία οδεύει προς την σωστή κατεύθυνση αλλά είναι ανεπαρκή σε ορισμένα σημεία. Αυτή τη στιγμή το σημαντικό είναι να διαπιστώσουμε σε τι δύσκολη περίοδο ζούμε στην Ευρώπη Σίγουρα πρέπει να περιορίσουμε τις μη απαραίτητες τα αλλά όχι με τέτοιο τρόπο που να κάνουμε περικοπές για χάρη των περικοπών. Πρέπει να είναι στόχο προσιλωμένες περικοπές να ευνοήσουμε την ανάπτυξη. Αν θέλουμε ανάπτυξη στην ευρωπαϊκή οικονομία, πρέπει να επενδύσουμε. Να επενδύσουμε στην έρευνα, στην έρευνα και ανάπτυξη, την καινοτομία, την εκπαίδευση. Αυτή είναι η βάση επί της οποίας μπορούμε να οικοδομήσουμε νέου τύπου ανάπτυξη στην Ευρώπη. Πολύ σημαντικό λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις στους τομείς που προανέφερα και φυσικά μπορούμε να περικόψουμε τα μη απαραίτητα αλλού, αλλά εκπαίδευση, καινοτομία, έρευνα τα χρειαζόμαστε αν πρόκειται να σταθεροποιήσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Καμίνσκι. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ, όπως ε, και όλοι οι Πολωνοί ε, της ομάδας ε, μεταρρυθμιστών και συντηρητικών ψήφισα διαφορετικό τρόπο. Ε, βέβαια, ε, αντιλαμβάνομαι τα επιχείρηματα αυτή που μιλούν για ανάγκη οικονομία και καταπολέμηση τη γραφειοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ αξιέπαινε αυτά τα συνθήματα και καλό είναι να τα υποστηρίξουμε. Αλλά θα πρέπει να ξεχνάμε ταυτόχρονα ότι οι περικοπές του ευρωπαϊκού προπολογισμού θα πλήξουν κυρίως τις νέε χώρες μέλη τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτές που κατεξοχήν χρειάζονται την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να κερδίσουν ε, το, ε, να κερδίσουν το χαμένο οικονομικό και πολιτιστικό έδαφος σε σχέση με τις πλούσιες παλιέ παλιές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς ε, ήδη από τι αρχέ τη δεκαετία του 1990 μόνο ανοίξαμε την αγορά μας και δεν προστατεύσαμε την αγορά μας κατά των Ολλανδικών, Βρετανικών και άλλων επιχειρήσεων που εποφελούνται από την πολωνική αγορά και τις διατάξεις. Σήμερα οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν, έχουν δικαίωμα να έχουν απαιτήσει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να βοηθεί και όχι να σταματήσει να βοηθεί. Γι' αυτό όλοι οι Πολωνοί της ομάδας ψήφισαν υπέρ αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ κύριε Καμίνσκι. Το λόγο έχει η κυρία Γιάτεν Μάκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ψήφισα υπέρ του παγώματος ε, του κοινοτικού προϋπολογισμού και είμαι υπέρ των περικοπών και της εξοικονόμησης ε, σε κοινοτικά κονδύλια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη ζουν με δάνεια ουσιαστικά και είναι υπερχρεωμένα. Θα πρέπει να επιτείνουμε τη χρέωση προκειμένου να ενισχύσουμε τον κοινοτικό προπολογισμό. Συνεχίζονται οι σημαντικέ και δραστικέ περικοπέ στου εθνικού προπολογισμού. Γι' αυτό αντίστοιχε εξοικονομήσει θα πρέπει να κάνει ο κοινοτικό προπολογισμό για να δώσει το καλό παράδειγμα. Θα πρέπει φυσικά να είμαστε καινοτόμοι και να βρούμε τρόπους ε, για εξοικονομήσει κονδυλίων. Δεν μπορούμε να επιτάσσουμε στα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν λιτότητα και να κάνουν περικοπές, ε, ενώ εμείς ε, να μην κάνουμε αντίστοιχε περικοπές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να βρούμε τομείς στους οποίους μπορούμε να επιβάλλουμε κάποιες οικονομίες. Όπως είπαμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να βρούμε κάποιους ευαίσθητους τομείς στους οποίους να πραγματοποιήσουμε οι Απ' την άλλη πλευρά θα πρέπει να επενδύσουμε στην ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στην επόμενη έκθεση. Μπορώ να υποστηρίξω γενικά τα μέτρα που ευνοούν την διαμεθοριακή συνεργασία σε, το σε τομείς αστικού δικαίου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω αυτό το ψήφισμα για την νομική κατάρτιση. Υπάρχουν ήδη μια σειρά πρωτοβουλίε που έχουν στόχο να λύσουν τα διαμεθοριακά νομικά προβλήματα. Άρα θα έχουμε επικάλυψη με πρωτοβουλίε που ήδη υπάρχουν. Επιπλέον η πρόταση αυτή για τη δημιουργία ενό ε, δικτύου έρασμο για του ε, δικαστέ είναι απόλυτα μη χρήσιμη και σπατάλη δεν σεβόμαστε έτσι την αρχή της επικουρικότητας, διότι τα νομικά συστήματα είναι σαφώς εθνικά ζητήματα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει εναρμόνιση ή συγκεντρω... Ε, συγκεντρωτισμό σε τέτοια θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Καμίνσκι. Κύριε Πρόεδρε, εγώ ε, ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος γιατί θεωρώ ότι ο ρόλος ε, και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των θεσμικών οργάνων είναι να βοηθήσουμε τους πολίτες. Εγώ είμαι υπέρμαχο φυσικά διαφοροποιημένη Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε διαφορετικέ ένωμε τάξει. Κάθε χώρα με διαφορετικό τρόπο προστατεύει του πολίτε, αλλά ταυτόχρονα είμαστε υπέρ των διαπροσωπικών σχέσεων και επαφών, υπέρ των οικονομικών επαφών μεταξύ των πολιτών διαφόρων χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θα πρέπει να εξοικειωθούμε περισσότερα με τα διάφορα νομικά συστήματα που θα ισχύσουν σε Ευρωπαίους πολίτες που διακινούνται όλο και περισσότερο, που ταξιδεύουν, που έχουν ε, σπουδές, παρακολουθούν σπουδές ή έχουν οικονομικές δραστηριότητες σε άλλες χώρες. Φυσικά, ε, στα πλαίσια της, ε, του κοινού νου και της ορθής λογικής χρειάζεται σημαντικός συντονισμός σε τέτοια θέματα. Σας ευχαριστώ. Προχωράμε τώρα στην επόμενη έκθεση. για την παιδική εργασία στον τομέα του κακάου. Το λόγο έχει η κυρία Μακλάρκιν. Συνάδελφοι, η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού καθιστά σαφή την ε, σημασία της εκπαίδευσης. Ιδίω ε, πρέπει να είναι υποχρεωτική και δωρεάν η εγκύκλια εκπαίδευση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την ανάπτυξη των νέων, ούτω ώστε να γίνουν υπεύθυνοι ενήλικε που να παίξουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία. Είναι πολύ επίγον λοιπόν να βοηθήσουμε την αντιμετώπιση του προβλήματος που είναι τα 250 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο που συνεχίζουν να εργάζονται ενώ δεν θα έπρεπε. Από τη φύση της η καλλιέργεια κακάου που μπορεί να είναι οικογενειακή επιχείρηση και θέλει πολλή εργασία. Στη Δυτική Αφρική καλλιεργείται το 70% της ε, παγκόσμιας, ε, του παγκοσμίου κακάου. Και αυτό βεβαίως ε, έχει να κάνει και με τι συνεχιζόμενες συγκρούσει στην περιοχή. Είναι δύσκολο να αλλάξει η κατάσταση. Αναγνωρίζω ότι υπάρχουν εργασίε που μπορεί να είναι αποδεκτό για τα παιδιά να συμμετέχουν εφόσον δεν του θερούμε τη δυνατότητα εκπαίδευση. Αλλά η καλλιέργεια κακάου είναι μεγάλο πρόβλημα για τα παιδιά γιατί του αφαιρεί τη δυνατότητα εκπαίδευση. Στηρίζω λοιπόν το ψήφισμα που εγκρίναμε για να είμαστε κατά τη υποχρεωτική καταναγκαστική εργασία παιδιών στον τομέα της ε, καλλιέργειας κακάο. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Τζανόνι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. 215 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο ε, δουλεύουν. 150 εκατομμύρια ε, είναι αυτά τα, παιδιά τα οποία έχουν ηλικία κάτω των 15 ετών και μάλιστα ε, δουλεύουν σε ιδιαίτερα επικίνδυνες εργασίες. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία δεν μπορούμε πλέον να ανεχτούμε. Εγώ υπερψήφισα την έκθεση για την παιδική εργασία στον τομέα του κακάου, γιατί πρέπει να είναι πολύ σημαντικό ο ρόλο που θα παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η νέα μορφή σκλαβιάς. Θα πρέπει στι εμπορικέ τη συμφωνίε, η Ευρωπαϊκή Ένωση με τι χώρε αυτέ, κυρίω δε με χώρε τη Δυτικής Αφρική, όπω α πούμε η ακτή του <coughs> ελεφαντοστού, που είναι κύριες παραγωγή ε, του κακάου θα πρέπει να βάλει ιδιαίτερη ρήτρα για την απαγόρευση της ε, παιδικής εργασίας ή της υποχρεωτικής παιδικής εργασίας στον τομέα του κακάου. Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε πλέον ε, προϊόντα τα οποία αποτελούν, την, την, αποτελούν αποτέλεσμα παιδικής εργασίας και αυτό θα πρέπει να φαίνεται και στα προϊόντα τα οποία φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σουίνμπερν. Ευχαριστώ. Η παιδική εργασία σε οποιοδήποτε τομέα είναι κάτι που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσπαθήσει να καταργηθεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν θα πρέπει να υπογράφουμε εμπορικέ συμφωνίε με το Πακιστάν και δεν θα πρέπει να αγοράζουμε κακάο από περιοχέ που το κάνουν αυτό. Θα πρέπει να καταλάβουν δηλαδή οι χώρε αυτέ ότι θέλουν να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αναγκαίο να έχουν ένα μήνυμο με επίπεδο προδιαγραφών. 215 εκατομμύρια παιδιά εργάζονται στον κόσμο. Σκανδαλώδες αυτό τη σημερινή εποχή. Πρέπει να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε την εμπορική μας δύναμη για να απαλείψουμε αυτές τις καταχρήσεις. Η εκπαίδευση των παιδιών είναι πιο σημαντικό, όχι να δουλεύουν από τόσο μικρά. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να υπάρξει ανάπτυξη και μια οικονομία πιο ζωντανή και δυναμική στο μέλλον. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρομπέρτα Αντζελίλη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε πολύ συχνά αγνοούμε τον τρόπο και τις προϋποθέσεις και τους όρους με τους οποίους παράγονται κάποια προϊόντα που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Δεν γνωρίζουμε λοιπόν ότι σε μερικές περιπτώσεις τα προϊόντα αυτά ε, καλλιεργούνται ή παράγονται με τη δουλειά 252 ε, εκατομμυρίων παιδιά, εκ των οποίων πολλά έχουν ηλικία κάτω των 15 ετών και ε, δουλεύουν σε πολύ επικίνδυνες δραστηριότητες. Στην περίπτωση αυτή υπόκειται και το, το κακάο. Ε, είναι λοιπόν ευθύνη και αρμοδιότητα όλων των χωρών που συμμετέχουν στην διαδικασία αυτή, κυρίως δε ε, των χωρών παραγωγών που αρνούνται να δημοσιοποιήσουν τα οικονομικά τους στοιχεία. Ε, και σε συνεργασία με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας ε, ευελπιστώ ότι θα δημιουργηθεί ένας οργανισμός ελέγχου των αλυσίδων παραγωγής έτσι ώστε να καταπολεμηθούν οποιαδήποτε μορφή κατάχρησης της εργασίας των παιδιών και να υπάρχει ενιχνεσιμότητα τα αυτή στα ε, προϊόντα του κακάου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρέπο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε στήριξα την έκθεση αυτή γιατί, ε, στην, γιατί στην Ευρώπη ε, συχνά καταναλώνουμε σοκολάτα ή προϊόντα κακάο τα οποία έχουν παραχθεί μέσα από τη δουλειά των παιδιών, ε, των ανηλίκων στην Γκάνα ή αλλού. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς επίσης και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα πρέπει να επιβλέπει τις διαδικασίες παραγωγής στις χώρες αυτές και να διασφαλίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα καθιερώσει Εμπορικέ εμπορικές σχέσεις με χώρες όπου είναι καθιερωμένη η παιδική εργασία. Ο τομέας του ε, κακάο ε, είναι ένα σημαντικό ε, στοιχείο που πρέπει να μας οδηγήσει σε νέα συμπεράσματα και βεβαίως δεν είναι μονάχα οι ευρωπαϊκές εταιρείες οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το ζήτημα. Είμαστε μια κοινότητα αξιών και δεν είναι δυνατόν να δεχόμαστε την χρήση παιδικής εργασίας στην παραγωγή και την συγκομιδή του κακάου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρέπο, η κυρία Ντότζ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Γύρω στις 250 εκατομμύρια ε, συγγνώμη, 250.000 παιδιά εργάζονται στι ε, καλλιέργειες κακάου στη Δυτική Αφρική. Τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει κάποιες προόδοι, πρωτοβουλίε για να αντιμετωπίσουμε τι μορφές μορφέ παιδικής εργασίας, αλλά πολλά πρέπει ακόμη να γίνουν. Η ακτή του εξάγει περίπου το μισό κακάο που εξάγεται στον, στον πλανήτη. Η χώρα αυτή ε, χυμάζεται από χρόνια εμφυλίου πολέμου και ακραία φτώχεια. Οι καλλιέργειες κακάου λοιπόν καλλιεργούνται από τα μέλη της οικογένειας συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών για να μειωθεί το εργατικό κόστος. Πιστεύω λοιπόν ότι ο μόνος τρόπος να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος παιδικής εργασίας είναι να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια αυτή. Είναι ο μόνος τρόπος ώστε χώρες όπως η φαντοστού να προοδεύσουν, να υπάρξουν δρόμοι, νοσοκομεία και κυρίως σχολεία για να μπορέσουν και τα παιδιά και οι γονείς τους να έχουν μια δυνατότητα καλύτερου μέλλοντος. Ευχαριστώ. Μπασέσκου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος γιατί η εκμετάλλευση των παιδιών και χρήση της παιδικής εργασίας ε, στη γεωργία της Δυτικής Αφρικής είναι ένα εξοργιστικό φαινόμενο και μάλιστα δυστυχώς έχει τεράστιες διαστάσεις. Η γενικευμένη φτώχεια και οι συγκρούσεις ε, έχουν επιδεινώσει την κατάσταση τα τελευταία χρόνια. Πέρυσι οι συγκρούσεις ε, στην ακτή του Ελεφανταστού οδήγησαν στον πλοκάρισμα 250.000 τόνων στην παραγωγή και μια αύξηση κατά 9% της τιμής ε, του κακάο στο χρηματιστήριο του Παρισιού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται από την Κάνα ή την ακτή του Ελεφαντοστού για τις εισαγωγές κακάο της. Βέβαια, ε, το εμπορικό στοιχείο δεν θα πρέπει να δημιουργήσει εμπόδιο στην συνεργασία μας με την Ίντερπολ στον τομέα αυτό, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το σωματεμπόριο και την εκμετάλλευση των παιδιών. Ε, θέλουμε να διευρύνουμε την ε, ιδέα του δίκαιου εμπορίου. Νομίζω ότι αυτό θα εξυπηρετήσει και τα συμφέροντα των παιδιών και των γονιών τους φυσικά. Ο κύριος Καμίνσκι. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ, φυσικά και τάχθηκα υπέρ του ψηφίσματος αυτού, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ κρίσιμες ε, στιγμές αυτές ε, στο κοινοβουλευτικό έργο. Γιατί παρά τις διαφορές μας που είναι πολλές φορές αισθητές ε, ενωνόμαστε σε σημαντικές αξίες και αρχές ξεπερνάμε αυτά τα χάσματα και ψηφίζουμε από κοινού σε ένα πρόβλημα όπως είναι ένα πρόβλημα που πραγματικά καλεί την εκδίκηση του ουρανού και την θεία οργή. Ε, Δυστυχώ εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο εξαναγκάζονται σε εργασία και ε, τη χάνουν εκμετάλλευση, ε, υπονομεύοντα ε, και το παρόν αλλά και το μέλλον τους. Αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη και εξορκιστική και χαίρομαι ιδιαίτερω που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολείται με το θέμα αυτό και χαίρομαι ιδιαίτερος που ασχολούμαστε με τέτοια θέματα γιατί θέλουμε να παρακολουθήσουμε τα κυκλώματα αυτά, με ποιο τρόπο φτάνουν τα προϊόντα αυτά στην ευρωπαϊκή αγορά γιατί εμείς είμαστε σημαντικός εισαγωγέ κακάο. Θα πρέπει λοιπόν να παρακολουθήσουμε, να ανοιχνεύσουμε όλα αυτά τα προϊόντα, να δούμε προϊόντα που αγοράζουμε στην Ένωση και τα πληρώνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες μήπως είναι παράνομα, μήπως είναι παράνομα από άποψη ε, διεθνούς δικαίου που φυσικά καταδικάζει τη χρήση της παιδικής εργασίας. Ευχαριστώ κύριε Καμίνσκι. Και τώρα η κυρία Σουίνμπαν για την επόμενη έκθεση. Όχι, συγγνώμη, Καμίνσκι. Ο κύριος Καμίνσκι για το διαβήτη. Φυσικά και τάχθηκα υπέρ της συμφωνίας αυτής για το κακάο. Με την συμφωνία αυτή αντικαθιστούμε την προηγούμενη συμφωνία ε, του 2001 και είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση αυτή η Διεθνή Συμφωνία για το κακάο. Βέβαια, απευθύνουμε έκκληση για τη διαφάνεια σε ό,τι αφορά την παραγωγή του κακάο. Το είπα και προηγουμένως. Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα με την παράνομη εκμετάλλευση παιδικής εργασίας στο κακάο. Μιλούμε επίσης ε, για κατάργηση των ε, εμπορικών φραγμών και για την ε, ευρεία πρόσβαση τέτοιων προϊόντων στην εσωτερική αγορά. Βέβαια, το κακάο είναι σημαντικό εξαγωγικό προϊόν φτωχών χωρών. Δεν θα πρέπει όμως ε, για, ε, για τη συγκομιδή κακάο να εκμεταλλεύονται οι χώρες αυτές τα παιδιά. Θέλουμε να εισάγουμε κακάο από τις φτωχές χώρες, να υποστηρίξουμε την ανάπτυξή τους, αλλά όχι πάση θυσία και όχι εις βάρος των παιδιών. Ναι, προφανώ έγινε ένα λάθο. Εγώ εδώ στην οθόνη είδα το όνομα τη κυρία Βίνμπορν, αλλά μίλησε ο κύριο Καμίνσκι. Η κυρία Βίνμπορν θα μιλήσει μετά από τον κύριο Τάκουλα. Πρώτα. Πρώτο συνάδελφο Τάκουλα. Πρόεδρε, ζήτησα το λόγο για την προηγούμενη έκθεση. Αλλά το θέμα είναι το ίδιο. Είναι σημαντικό θέμα πρέπει να υποστηρίξουμε τις αξίες μας και μία κεντρική αξία μας είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και τα ανθρώπινα δικαιώματα συμπεριλαμβάνουν τα δικαιώματα των παιδιών. Πρέπει να αποδώσουμε λοιπόν την αναγκαία προσοχή στο θέμα αυτό, ούτως ώστε ανεξάρτητα από τις συνθήκες τα παιδιά δεν χρειάζεται να εκτίθενται σε τέτοιου τύπου εργασία, αλλά αντίθετα διασφαλίζουμε την ανάπτυξη των παιδιών και επίσης λαμβάνουμε υπόψη τις ψυχολογικές και ε, γνωσιακές ανάγκες ανάπτυξης των παιδιών και κινητικές επίσης. Πρέπει λοιπόν να είμαστε κάθετα κατά της παιδικής εργασίας. Όταν συνάπτουμε εμπορικές συμφωνίες με τις χώρες αυτές, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι εταίροι μας δεν εκμεταλλεύονται τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο. Και γι' αυτό Πρέπει να εμποδίζουμε οποιασδήποτε εξοικονομήσει σε βάρο των παιδιών. Τα, δικαιώματα έχουν, τα παιδιά έχουν δικαίωμα ε, σε παιδική εργασία. Και τώρα η κυρία Σουίνμπερν. Ευχαριστώ. Η κατάργηση των εμπορικών φραγμών με τη βοήθεια άλλων των χωρών και του ιδιωτικού τομέα. Αυτό είναι ο τρόπο τον οποίο πρέπει να λειτουργεί η παγκόσμια αγορά. Πρέπει να διευκολύνουμε σε περισσότερου τομεί την δραστηριότητα αυτή. Θέλουμε κυρίως να υπάρξει περισσότερη ανάλυση, στατιστικά στοιχεία και μελέτες επιπτώσεων για τους λόγους των εμπορικών φραγμών στον τομέα αυτό. Ελπίζω έτσι να πάρουμε πιο σωστές αποφάσεις για να υπάρξει καλύτερη ρύθμιση της αγοράς αγαθών. Στόχος μας είναι να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία για κάθε προϊόν για να έχουμε έναν ιδιαίτερα εκλεπτισμένο μηχανισμό ούτως ώστε να μην εμποδίσουμε τη δραστηριότητα των παραγωγών και των καταναλωτών που προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε δραστηριότητα των παραγών αυτών με αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στο επόμενο ψήφισμα. Είναι το ψήφισμα για, για το διαβήτη και θα δώσω το λόγο πάλι στην κυρία Σουίνμπερν. Ευχαριστώ πολύ. 10% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποια στιγμή της ζωής του παρουσιάζει διαβήτη. Με τον γυράσκοντα πληθυσμό αυτό το ποσοστό θα αυξηθεί δραματικά τα επόμενα χρόνια. Ε, ε, υπάρχουν τύποι διαβήτη όπως ε, κάποιοι τύποι του τύπου Α που μπορούν να ιαθούν. Επίσης ο διαβήτης τύπου Β μπορεί να θεραπευτεί μέσα από καλύτερη ζωή, καλύτερες συνήθειες, άσκηση κτλ. Είναι σόφρον να αναλάβουμε μια κοινή δράση απέναντι στο θέμα αυτό και βεβαίως και σε όλες τις χώρες να υπάρξει ένα σύστημα πρώιμης διάγνωσης του διαβήτη. Αυτό μαζί με μια κοινή πολιτική αντιμετώπιση ε, και την έκδοση ε, κατευθυντηρίων γραμμών θα μπορέσει να βελτιώσει την κατάσταση. Ψήφισα ε, αυτό το ψήφισμα γιατί πιστεύω ότι θα είναι ωφέλιμη μια κοινή στρατηγική τη Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα αυτό ε, κυρίως ε, γιατί πρόκειται για μια ασθένεια η οποία βαραίνει πολύ τα ταμεία σε μια οικονομικά δύσκολη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ τώρα η κυρία Γιανακουδάκη. Ευχαριστώ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο περίπου 3 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από διαβήτη με άξερση της παχυσαρκίας και γύρωση του πληθυσμού, το κόστος του διαβήτη για το σύστημα υγείας ε, θα, ανέλθει, θα αυξηθεί κατά 10% στον ετήσιο προϋπολογισμό της υγείας. Αυτές είναι οι προβλέψεις. Και μάλιστα δεν είναι απομονωμένο το φαινόμενο ε, του Ηνωμένου Βασιλείου. Φαίνεται ότι κατά πάσα πιθανότητα ένας στους 10 πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, υποφέρουν από διαβήτη. Βέβαια η υγεία είναι εθνική αρμοδιότητα, αλλά πιστεύω ότι η ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών θα αποβεί σε όφελο όλων μας μια στρατηγική που βελτιώνει την, το συντονισμό, τη συνεργασία, ενισχύει την έρευνα και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, μας δίνει ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε την, την τεχνογνωσία και τους πόρους που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια επιδημία που αν συνεργαστούμε μπορούμε να την ελέγξουμε. Για όλου αυτού του λόγου, λοιπόν τάχθηκα υπέρ τη έκθεση. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Αντζελίλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι ανησυχητικά τα στοιχεία τα, αυτά τα οποία αφορούν ε, τον διαβήτη. Πρόκειται για πραγματική επιδημία ε, με παραπάνω από 300.000 θανάτους κάθε χρόνο. Μία χρόνια ασθένεια η οποία έχει αυξήσει τον τελευταίο καιρό τις ταπάνες υγείας από το 10% στο 26%. Μπορούμε να ε, αντιμετωπίσουμε την ασθένεια αυτή έστω και αν ξέρουμε ότι δεν είναι μεταδοτική αλλά ε, που είναι μια ασθένεια η οποία θα αυξηθεί ε, λόγω ε, εσφαλμένων τρόπων διαβίωσης και λόγω του γυράσκοντος πληθυσμού. Πρέπει λοιπόν να, ληφθούν, να αναλυφθούν δράσεις όσον αφορά την πρόληψη ας πούμε της παχυσαρχίας καθώς επίσης και εκστρατείες οι οποίες θα προωθούν τον υγιή τρόπο ζωής. Επίσης σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει η στρατηγική να είναι καινοτόμα, στοχευμένη ε, και ε, προοδευτική έτσι ώστε ε, να δοθούν και απαραίτητα χρήματα σε προγράμματα έρευνας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Αντζελίλη. Ο κύριος Ρέπο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ ψήφισα υπέρ της έκθεσης γιατί ο διαβήτης εκτός της προσωπικής οδύνης συνεπιφέρει μεγάλο κόστος και για την κοινωνία. Δυστυχώς ο διαβήτης ε, επεκτείνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια ο διαβήτης τύπου 2 σχετίζεται και με τον τρόπο ζωής. Γι' αυτό και θα πρέπει να έχουμε παρκείς πληροφορίες και για τα τρόφιμα και να δούμε ποια διατροφή ενδείκνεται για την καταπολέμηση την πρόληψη του διαβήτη. Η ετικετοθεσία στα τρόφιμα δεν θα πρέπει να είναι παραπλανητική για να μπορούν οι καταναλωτέ ε, να διαμορφώνουν περιστατωμένα τη γνώμη τους για να επιλέγουν το τρόφιμά τους. Ο διαβήτης ε, μπορεί να προληφθεί με τις σωστές διατροφικές συνήθειες και με σωματική άσκηση γιατί ε, η επιρροή του διαβήτη στην υγεία είναι πολύ σημαντική. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε έμφαση στην πρόληψη με κάθε μέσο και γι' αυτό τάχθηκα αναφανδόν υπέρ της έκθεσης. Ευχαριστούμε κύριε Ρέπο. Το λόγο έχει η κυρία Ντότζ. Ευχαριστώ. Τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι 2,9 εκατομμύρια στο Ηνωμένο έχουν διαγνωστεί με διαβήτη. Το στοιχείο αυτό συμπεριλαμβάνει και αυτούς που είναι στη δική μου εκλογική περιφέρεια Βόρεια Ιρλανδία 73,5 άτομα και φαίνεται ότι υπάρχουν και χιλιάδες που δεν έχουν ακόμη διαγνωστεί. Αυξάνεται λοιπόν στη Βόρεια Ιρλανδία, όπως παντού στην Ευρώπη, ο διαβήτης τα τελευταία 6 χρόνια. Στην εκλογική μου περιφέρεια, ο αριθμός των ατόμων με διαβήτη που έχουν διαγνωστεί έχει αυξηθεί περίπου 41% μια πρόσφατη μελέτη με τίτλο «Ο διαβήτης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας» ε, θεωρεί ότι πρέπει να δαπανηθούν 3,5 δισεκατομμύρια το χρόνο. Αυτό είναι πάνω από 9,6 εκατομμύρια τη μέρα για τη μετώπιση της ασθενείας αυτής. 100.000 ε, ε, άτομα διαγνώσκονται με διαβήτη κάθε χρόνο στον Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη πίεση στα κονδύλια. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο ενεργοί στην αντιμετώπιση μέσω ε, εκπαίδευσης και αύξησης της συνειδητοποίησης και πρέπει να βελτιώσουμε την ε, διατροφή των ατόμων και την άσκηση. Ευχαριστώ. Μπασέσκου. Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης γιατί νομίζω ότι η καταπολέμηση του διαβήτη πρέπει να ενισχυθεί με όλα τα δυνατά μέσα. Πιστεύω κυρίως στην πρόληψη μέχρι το 2030 πάνω από 16% των πολιτών της Ευρώπης θα θυγούν από την ασθένεια αυτή. Πρέπει λοιπόν να ενημερώσουμε τον πληθυσμό για το θέμα αυτό, να τον εκπαιδεύσουμε δυστυχώς. Ο διαβήτης δεν μπορεί να θεραπευθεί, αλλά υπάρχουν ε, τρόποι πρόληψης. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επενδύσει περισσότερο στην ε, προώθηση του αθλητισμού, της αθλητικής δραστηριότητας, και να ενθαρρύνει έναν υγιή τρόπο ζωής. Και επίσης πρέπει να γίνεται έγκαιρη διάγνωση του διαβήτη και τύπου 1 και τύπου 2. Αυτό θα μπορούσε να διασφαλίσει την κατάλληλη αντιμετώπιση της ασθένειας και να μειώσει τις δαπάνες που προκύπτουν λόγω των ε, επιπλοκών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τάνοκ. Εγώ είμαι υπέρ ε, της έκθεσης αυτής, γιατί βεβαίως η υγεία είναι κυρίως εθνικό θέμα, αλλά οι περιορισμένες προτάσεις που τίθενται θα έχουν θετική επίπτωση στον τομέα της έρευνας για τον διαβήτη. Περίπου 10% του πληθυσμού της ε, Ένωσης θίγεται και είναι πάνω από 10% των δαπανών στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή ε, γυράσκει ο πληθυσμός θα αυξηθεί η δαπάνη αυτή. Πρέπει να υπάρξει ομοφωνία στον τομέα της δημόσιας υγείας μεταξύ των κρατών μελών για να υπάρξει ένας μηχανισμός που να ε, ενημερώνει για τις βέλτιστες πρακτικές για να προλάβουμε, να διαγνώσουμε και να παρακολουθήσουμε. Πρέπει να συνεχιστεί η χρηματοδότηση της έρευνας μέσω του προγράμματος πλαισίου ως ε, γιατρός και ως μεσήλικας και κάπως ε, υπέρβαρος. Ε, κινδυνεύω να πάθω διαβήτη 2 που δυστυχώς ήταν η αιτία θανάτου του ε, παππού μου. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος αυτού, γιατί είναι πολύ σημαντικό και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να μη φυστούμε προσπαθειών προκειμένου να προλάβουμε την, το διαβήτη ή να περιορίσουμε την εμφάνισή του. Έχει φτάσει σε διαστάσεις επιδημίας δυστυχώς. Υπάρχει μια έξαρση της ασθένειας αυτής. Βέβαια, περισσότερο μιλούμε για το διαβήτη τύπου 2, που οφείλεται σε αλλαγή του τρόπου ζωής. Σίγουρα η διατροφή και η σωματική άσκηση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υγεία του ανθρώπου. Τα θέματα υγείας βέβαια είναι σε μεγάλο βαθμό εθνική αρμοδιότητα. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να δείξουμε κάποια ευαισθησία για τους κινδύνους της υγείας και να θαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να φροντίσουν ότι, ώστε ήδη από το σχολείο να ενημερώνονται οι μαθητές για τα θετικά αποτελέσματα μιας υγιεινής διατροφής και ενός υγιεινού τρόπου ζωή. Θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε να προλάβουμε αυτή την έξαρση του διαβήτη τύπου 2. Ο κύριος Καμίνσκι, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, 10% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι άνθρωποι που πάσχουν από διαβήτη, που δίνουν τη μάχη τους κατά του διαβίτη. Και με τις αλλαγές στον τρόπο ζωής, με την πολιτιστική, ε, ε, πολιτιστική ανάπτυξη, αλλά και με τη γύραση του ευρωπαϊκού πληθυσμού, το πρόβλημα του διαβήτη θα αφορά όλο και περισσότερους συμπολίτε μας δυστυχώς. Γι' αυτό και υπερψήφισα ε, την έκθεση αυτή, το ψήφισμα αυτό, γιατί θεωρώ ότι η κλίμακα του προβλήματος του διαβήτη είναι τόσο μεγάλη πια σήμερα, έχει ξεπεράσει τα εθνικά σύνορα, γι' αυτό και θα πρέπει ε, να συνενώσουμε πανευρωπαϊκά τις προσπάθειές μας για να καταπολεμήσουμε αυτό το πρόβλημα. Να δώσουμε έμφαση στην υγιεινή διατροφή, στο υγιεινό τρόπο ζωής και να ενισχύσουμε φυσικά και τις ε, ιατρικές εξετάσεις ε, για πρόορη διάγνωση του διαβήτη. Χαίρομαι ειλικρινά γιατί με συντριπτική πραγματικά πλειοψηφία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε το ψήφισμα αυτό. Σας ευχαριστώ κύριε Καμίνης και ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, είναι σαφές ότι είναι πολύ σωστό που μιλάμε τώρα για αυτό το τόσο σημαντικό ε, ζήτημα. Θα πρέπει να βρούμε καλύτερους τρόπους αντιμετώπισης της ασθένειας και ακόμα καλύτερα τρόπους ε, να προλάβουμε την ασθένεια αυτή. Ε, πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι 90% ε, ε, των ιατρικών δαπανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούν να καταπολεμήσουν ασθένειες και μονάχα 3% του ιατρικού προϋπολογισμού αφορά την έρευνα. Γι' αυτό λοιπόν θα συμφωνήσω απολύτως με την Κέντ Σουίνμπορν η οποία λέει ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε την έρευνα όσον αφορά την πρόληψη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ θέλουν να αλλάξουν την, τον τρόπο ζωής τους ε, και μπορούν, μπορούμε σε αυτόν τον τομέα να κάνουμε έρευνα. Ε, είναι, επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε και την σημασία της αθλητικής ε, δραστηριότητας και κυρίως στα πλαίσια του κοινωνικού ταμείου θα πρέπει να βρούμε και μια ειδική αναφορά στις αθλητικές δραστηριότητες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κέλλη και περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο έκθεση σχετικά με τη διεύρυνση για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ευχαριστώ. Χαιρετίζω τα θετικά που υπόθηκαν στην έκθεση για την διεύρυνση με την μου Και άλλες χώρες ε, ένταξης όπως η Σερβία που έγινε δεκτή την προηγούμενη εβδομάδα ως ε, υποψήφια χώρα θα μπορούσαν να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Μακεδονίας πώς έχει συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δύο χώρε είχαν ε, παρόμοια προβλήματα στο παρελθόν. Πρέπει να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και του πληθυσμού του και τι συνεχιζόμενε ε, διαμάχε με του ε, γείτονέ του. Η διαμάχη με την Ελλάδα για το θέμα τη ονομασία δεν θα πρέπει να συγκριθεί με την διαμάχη Βελιγραδίου και Πρίστινα. Αλλά ο τρόπο που αντιμετωπίζει η Μακεδονία για να αντιμετωπίσει αυτή τη διαμάχη μπορεί να είναι μια καλή αρχή και για άλλε χώρε, συμπεριλαμβανομένη και τη Σερβία, ω πρότυπο για τη συμπεριφορά του τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Αντωνιώτση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ πήγα προσωπικά στην Μακεδονία στις τελευταίες προεδρικές εκλογές ως απεσταλμένος από την πολιτική ομάδα του του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ε, και είχα την ευκαιρία να συνειδηθώ και με τον Πρωθυπουργό Γκρούεσκι. Ε, επομένως ε, είδα ότι όχι μονάχα τα θεσμικά όργανα αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες θέλουν οπωσδήποτε ε, να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε για ακόμα πολύ χρόνο τις διαπραγματεύσεις οι οποίες σταμάτησαν κάποια στιγμή και που θα πρέπει να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις αυτές. Η έκθεση του 2000 έκθεση προόδου του 2011 που υπέβαλε η Επιτροπή δείχνει ότι για τρίτη συνεχόμενη χρόνια η ε, δημοκρατία της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας ε, κατάφερε να προχωρήσει και να προσεγγίσει τα ευρωπαϊκά κριτήρια όσον αφορά την οικονομία της αγοράς ε, και επομένως θα πρέπει να ξεπεραστούν τα πολιτικά, οι πολιτικές δεσμεύσεις που ακόμα την κυρώνουν και επομένως να προχωρήσουμε τις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, είναι πραγματικά ε, πολύ κρίμα που εξαιτία της διαμάχης για την ονομασία καθυστερεί η διεύρυνση και προς τη Μακεδονία και αναχαιτίζει την ε, ταξιακή διαδικασία της χώρας αυτής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποσχέθηκε προσχώρηση σε όλες τις χώρες των Βαλκανίων και η Μακεδονία ήταν από τις πρώτες χώρες που έλαβαν το χαρακτηρισμό της υποψήφιας χώρας ε, για ένταξη. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις ε, φιλοευρωπαϊκές βλέψεις αυτής της χώρας. Για τρία συνεχή χρόνια η σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, προς το Συμβούλιο ήταν η έναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξης, παρόλο που το Συμβούλιο δεν συμφώνησε. Ε, δεν πρέπει να επιβάλλεται ήδη μια ε, λεκτική λογοκρισία και δεν ε, χρησιμοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση όρος Μακεδονία, κάτι που δεν ισχύει για τα Ηνωμένα Έθνη που χρησιμοποιείται η ονομασία εκεί. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε καμιά χώρα πίσω, να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας, γιατί διαφορετικά θα δικηβεύσουμε την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόοδος της Μακεδονίας θα εξαρτηθεί φυσικά από την ίδια τη χώρα. Αλλά σίγουρα δεν θα πρέπει να κλείσουμε τι πύλε τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ τη χώρα αυτή μόνο και μόνο εξαιτία τη διαμάχη του ονόματο. Ο κ. Κυρίλο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι πρόοδοι της πρώην Ιουκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας καταδεικνύουν την ισχυρή θέληση της χώρας αυτής να ε, μπει πλέον και να συμμετάσχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, είναι σε στρατηγικό σημείο ε, των Βαλκανίων, έχει ενστερνιστεί πολλές ευρωπαϊκές διαδικασίες και επομένως θεωρούμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Όσον αφορά το εκανθόδε ζήτημα της αποκέντρωσης της γραφειοκρατίας, ε, ήδη τα πρώτα σημάδια είναι θετικά και μας αφήνουν καλές ελπίδες για το μέλλον. Παραμένουν βεβαίως και στοιχεία ιδιαίτερα ανησυχητικά όσον αφορά τη διαφθορά, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διαφορά και την διαπλοκή μάλλον των μέσων ενημέρωσης. Ε, ε, βεβαίως θα πρέπει να δυναμωθούν τα κίνητρα όσον αφορά τον εκδημοκρατισμό της χώρας. Πιστεύω ότι σε μια ισχυρή και πιστεύω σε μια ισχυρή και διευρυμένη Ευρώπη, γι' αυτό ψήφισα αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πυρίλο. Στο Γιάννοφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για πρώτη φορά από τότε που έγινε Ευρωβουλευτής ψηφίζω κατά μιας έκθεσης σχετικά με τη διεύρυνση μιας χώρας, συγκεκριμένα της πρώην Ιουκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας. Στο παρελθόν υπερψήφιζε γιατί θεωρούσε ότι έτσι θα παροτρύναμε την Μακεδονία να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις της. Πέντε χρόνια έχουν περάσει που είναι συνήθως ε, η προθεσμία που χρειάζεται μια χώρα ή μάλλον ε, το μισό της προθεσμίας που χρειάζεται μια χώρα για να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, δυστυχώς όμως στη Μακεδονία συνεχίζονται οι διώξει ε, κατά των ε, ε, Βουλγαρών όσων διεκδικούν την βουλγαρική εθνικό, εθνότητα. Υπάρχουν περιορισμοί και ω προ τη γλώσσα και στα μέσα μαζική ενημέρωση. Δεν πρόκειται να υποστηρίξω την ένταση μια χώρα που δεν πληρεί τα πολιτικά κριτήρια για την προσχώρησή τη. Δεν πρόκειται να υποστηρίξω μια χώρα που αντιμετωπίζει με τέτοιο τρόπο του υπηκόου τη γειτονική χώρα και που καταστρατηγεί την ελευθερία έκφραση και την ελευθεροτυπία. Ευχαριστώ η κυρία Μπασέσκου. Σας ευχαριστώ. Εγώ ψήφισα υπέρ της έκθεσης γιατί η σταθερότητα στα Βαλκάνια είναι πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα Σκόπια σημείωσαν κάποια πρόοδο ό,τι αφορά τι δημοκρατικέ μεταρρυθμίσει. Θα πρέπει όμω να συνεχιστούν αυτέ αδιαλείπτω, ιδιαίτερα στον δικαστικό τομέα ή στην καταπολέμηση τη διαφθορά. Ταυτόχρονα θα ήθελα να υποστηρίξω την ανάγκη για περισσότερη διαφάνεια των ε, δαπανών, των κρατικών δαπανών και τη χρηματοδότηση των ε, πολιτικών κομμάτων. Εκτιμώ τις προσπάθειες των μακεδονικών αρχών που θεωρούν ότι ο πλουραλισμός ε, και η πολιτισμικότητα είναι το χαρακτηριστικό της χώρας. Για παράδειγμα, η ρωμαϊκή εθνότητα αναγνωρίζεται και τη χάνει προστασίας. Επίσης, οι ΡΟΜ καλύπτονται από το εκπαιδευτικό σύστημα και εκπροσωπούνται στη δημόσια διοίκηση. Θα πρέπει όμω να συνεχιστούν οι προσπάθειε για να βελτιωθεί η κατάσταση αυτών των κοινοτήτων. Πρόεδρε, η ομάδα μου υποστήριξε την έκθεση αυτή. Καλούμε το Συμβούλιο να βεβαιώσει την έκκληση τη Επιτροπή για κατά προτεραιότητα ε, ημερομηνία για διαπραγματεύσει, για έναρξη των διαπραγματεύσεων. Η συνέχιση τη αρνησικυρία τη Ελλάδα έχει κρατήσει υπερβολικά πολύ. Διμερεί θέματα δεν θα πρέπει να είναι εμπόδιο στην περαιτέρω ένταξη τη Μακεδονία στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπω έχει γίνει από τότε που δόθηκε καθεστώ υποψηφίου στη χώρα από το 2005. Υπό τον ε, Πρωθυπουργό Γκρουεύσκη έχει υπάρξει μεγάλη πρόοδο στην ε, εθνική συμφιλίωση, την αποκέντρωση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημόσια δίκηση. Ο υπεύθυνο και μετρημένο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι εθνοτικέ εντάσει μεταξύ των Σλάβων και των Αλβανών στη χώρα είναι απόδειξη της πρόοδου και η πρόσφατη απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου κατά της, του βέτο της Ελλάδας για την ένταξη της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ πρέπει να γίνουν αντικείμενο σεβασμού από όλη την Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Τάνοκ. Ο κύριος Μπίλαν. Ευχαριστώ. Η διεύρυνση και προς τα Βαλκάνια αποτελεί ένα επιπλέον στάδιο στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η, η δημοκρατία της Μακεδονίας είναι ήδη σημαντικός κοντινός εταίρος Ευρωπαϊκής Ένωσης στα οικονομικά θέματα. Ο άμεσος προσδιορισμός ημερομηνία έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα στη σχέση μας με τη χώρα αυτή. Αναγνωρίζω επίση τη φιλοευρωπαϊκή πολιτική των Σκοπίων καθώ και τι ευρωατλαντικέ τη βλέψεις όπω φαίνεται από την υποψηφιότητα τη χώρα αυτή για το ΝΑΤΟ. Τα θέματα τη Ευρωπαϊκή ασφάλεια θα πρέπει να συμβαδίζουν με την ιδέα της διεύρυνση. Αξιοσημείωτη είναι επίση η οικονομική πρόοδο τη Μακεδονία, όπω φαίνεται στην έκθεση τη Παγκόσμια Τράπεζα, που τη φέρνει τρίτη χώρα σε ό,τι αφορά την επιτυχία κανονιστικών μεταρρυθμίσεων την τελευταία πενταετία. Επιτυχημένη ήταν και η στρατηγική καταπολέμηση της διαφθοράς, όπως φάνηκε και από την ε, βελτίωση της θέσης ε, της χώρας αυτής στην κατάταξη της διεθνούς διαφάνειας. Πιστεύω στο ε, οικονομικό δυναμικό αυτής της χώρας και στην σταθεροποίηση της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης που θα αποτελέσει και την ισχύ της διαπραγματευτικές διαδικασίες. Ευχαριστούμε κύριε Μπιέλαν, ο κύριος Καμίσκι. Κύριε Πρόεδρε, τα Βαλκάνια για πολλά χρόνια ήταν η πυρητιδακοποθήκη της Ευρώπης και ένα σημείο, μια περιοχή που επικρατούσε ανασφάλεια. Σήμερα χαιρετίζουμε και επικρατούμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση το γεγονός ότι όλο και περισσότερες χώρες των Βαλκανίων δηλώνουν και μάλιστα ειλικρινά τις φιλοενταξιακές τους προσδοκίες και τις βλέψεις τους για ένταξη σε μια κοινότητα που ε, δημιουργεί μια ένωση άνευ προηγουμένου και αποτελεί ένα χώρο οικονομικής ε, ανάπτυξης, ευημερίας και πρώτα απ' όλα ειρήνης. Χώρες που βίωσαν ε, τέτοια εμβόλυμες καταστάσεις επιτέλους ζητούν ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι υπέρ της ενταξιακής προσδοκίας της Μακεδονίας και απευθύνω έκκληση προς τους Έλληνες να μην επιμείνουν σε αυτό το πρόβλημα της, της ονομασίας. Νομίζω ότι στενές σοβινιστικές προσεγγίσεις δεν έχουν τη θέση τους εδώ. Θα πρέπει όλοι με κατανόηση και με φιλικό πνεύμα ε, και αμοιβαία κατανόηση να ζήσουμε αρμονικά και από κοινού στην Ευρωπαϊκή μας Ήπειρο. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στην έκθεση για την Ισλανδία. Κυρία Σουίνμπερν. Ευχαριστώ συζητώντας την ε, διαδικασία διεύρυνση με την Ισλανδία, είναι πολύ δύσκολο να το κάνουμε μόνο σε τεχνικό επίπεδο με βάση τα κριτήρια της Κοπενχάγης και το κεκτημένο, γιατί είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση από τις χώρες που μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την πτώση του τείχους του Βερολίνου και την ε, κατάρρευση του Ανατολικού Συνασπισμού. Πρέπει οπωσδήποτε να διαπιστώσουμε εάν η Ισλανδία πληρεί όλα τα κριτήρια. Για παράδειγμα, στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ούτως ώστε η τροποποιημένη, η μεταρρυθμισμένη Ισλανδική ε, οικονομία και ο τραπεζικό τομέα πληρούν όλα τα κριτήρια. Γιατί υπάρχουν πολλέ ανησυχίε για το θέμα αυτό στον Άνω Βασίλειο. Γιατί πολλά άτομα και πολλέ τοπικέ αρχέ έχασαν σημαντικά ποσά λόγω το αποτυχημένο ρυθμιστικό σύστημα του τραπεζικού τομέα στην Ισλανδία. Υπάρχει αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και χωρισμένα. Πρέπει να διασφαλίσουμε την επίλυση του ζητήματο αυτού όσο το δυνατόν πιο σύντομα να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για να μην επαναληφθεί. Ευχαριστώ. Χάναν. Ευχαριστώ. Υπήρξε πολύ μνησικακία στην ε, Ισλανδία ε, όταν κατέρευσε η Ισλανδία. Ήρθαν και μου είπαν, κοίταξε Χάναν, πώς πάνε τώρα οι Ισλανδοί σου. Αυτό παθαίνει όταν είσαι εκτός Ευρώπης. Ποιος όμως τώρα έχει το, την τελευταία λέξη. Η Ισλανδία μπόρεσε να υποτιμήσει, έτσι μπόρεσε να κάνει εξαγωγέ και έχει περισσότερη ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή την ζηλεύουν οι χώρες της Ευρωζώνης. Επειδή δεν έκανε αυτό το τρομερό λάθος να αναλάβει τα κακά χρέη ιδιωτικών οργανισμών, μόλι λυθεί το θέμα αυτό, θα έχει μια θαυμάσια οικονομική ανάπτυξη. 67% των Ισλανδών είναι κατά τώρα τη ένταξη στην Ένωση και καταλαβαίνουν τι θα σημαίνει αυτό. Θα του πάρουν του πόρου του, θα διάσουν οι θάλασσέ του και η δημοκρατία του, η παλιότερη δημοκρατία στον κόσμο θα γίνει χωρί περιεχόμενο. Είναι ιδιαίτερα ευφύοι άτομα επειδή έχουν αντιμετωπίσει πολύ δύσκολε συνθήκε εδώ και αιώνε, δεν θα κάνουν αυτό το λάθος. Ευχαριστώ η κυρία Γιανακουδάκη. Μου κατά του ψηφίσματος. Όχι επειδή νομίζω ότι δεν πρέπει να ενταχθεί η Ισλανδία, αλλά γιατί το ψήφισμα λέει ότι τα χρήματα που χρεώνει, που χρωστάει η Landsbanki της Ισλανδίας μετά την κατάρρευση του ISEV δεν πρέπει να είναι εμπόδιο στην ένταξη. Ω συντηρητική ευρωβουλευτή για το Λονδίνο δεν μπορώ να συμφωνήσω με τέτοιου όρου. Οι τοπικέ αρχέ στο Λονδίνο υποφέρουν τρομερές περικοπές λόγω 13 ετών ε, δαπανηρού και σπάταλου εργατικού καθεστώτος. Έξι τοπικές αρχές είχαν ε, επενδύσει 120 εκατομμύρια στο ISEV. Το μετρό του Λονδίνου 40 εκατομμύρια. Η, το, η αστυνομία του Λονδίνου 30 εκατομμύρια. Χάθηκαν όλα αυτά τα λεφτά από τότε που κατέρευσαν τον Οκτώβριο του 2008 οι Ισλανδικές τράπεζες. Η κυβέρνηση της Ισλανδίας αποφεύγει τις νομικές της υποχρεώσεις, τις νόμιμες υποχρεώσεις να πληρώσει ένα μίνιμουμ αποζημίωση στους Βρετανούς δανειστές της. Η Θάτσορ κάποτε είπε «Θέλουμε να μας επιστραφούν τα χρήματά μας». Αυτό ζητάμε τώρα από την Ισλανδία. Μέχρι να μας πληρώσουν δεν μπορώ να υποστηρίξω την ένταξή τους. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Ρέπο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε σε αυτήν την κατάσταση κρίσης και εμείς ε, οι πολιτικοί καμιά φορά ξεχνάμε πόσο η ευζοία και η σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει βοηθήσει τα, ε, τους πολίτες της ε, να βιώνει η οικονομία της Ισλανδίας και είναι καλό αυτό γιατί πρόκειται για μια χώρα με βαθιές δημοκρατικές ρίζες και παλιά δημοκρατική παράδοση. Ε, επίσης ε, πιστεύουμε ότι θα είναι ε, μια καλή στρατηγική προώθηση προς την Αρκτική, κυρίως όσον αφορά και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ήδη αυτή τη στιγμή καλύπτει η Ισλανδία τα κριτήρια της Κοπενχάγης και επομένως από τώρα θα μπορούσε να είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως υπάρχουν θέματα όπως η φαλαινοθυρία, πούμε, η οποία δημιουργεί προβλήματα ε, και βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη για τις επιτυχίες της κάθε χώρας ε, μπορούμε να πούμε ότι ήδη η Ισλανδία θα μπορούσε να γίνει μέλος. Ευχαριστώ πολύ. Κάμπελ. Uh, Πρόεδρε, καταψήφισα την ένταξη της Ισλανδίας γιατί νομίζω ότι όπως και τα δύο τρίτα των ε, Ισλανδών σε μια δημοσκόπηση τον τελευταίο μήνα η Ισλανδία θα ήταν τρελή να μπει στην Ένωση. Τρέλα θα ήταν αυτό, θα καταστρέψει την κύρια οικονομική της δραστηριότητα την αλληλεία μέσω της ε, καταστροφικής κοινή αλληλευτικής πολιτικής όπως κατέστρεψε εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σχεδόν όλοι οι αλληλείς έχουν χάσει τη δουλειά τους στη δική μου περιοχή. Και επίσης ε, γιατί θα έμπαιναν ε, στην Ευρωζώνη και να εγκαταλείψουν το νόμισμά τους που τους επιτρέπει να κάνουν εξαγωγές. Τρέλα γιατί θα είχαν όλη την κοινοτική γραφειοκρατία στην πλάτη τους η πρόβλεψη για την ε, αύξηση του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 0 φέτος, ενώ αυτοί έχουν 1,3. Γιατί λοιπόν να μην ε, βασιστούν ε, όμως οι προσπάθειες που κάνουμε να πάρουμε τα χρήματά μας μέσω της ΕΦΤΑ που πρότεινε να τα λάβουμε αυτά τα χρήματα. Στόχος των Ισλανδών είναι να παραμείνουν περήφανοι, ανεξάρτητοι και αυτόνομοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κυρία Ευχαριστώ. Στον Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει μια εκλογική περιφέρεια. Ή μάλλον ένα τμήμα του πληθυσμού είναι, θα μπορούσε να συμβουλεύσει του Ισλανδού να μείνουν έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν κάνει κανεί αίτηση να ενταχθεί σε οποιοδήποτε οργανισμό, πρέπει να αποδείξει σαφώ ότι πληρεί τα κριτήρια ότι δέχεσαι τους ε, κανόνες και τους ε, εφαρμόζεις. Ιδιαίτερα όσον αφορά το γάδο. Η Ισλανδία δεν έχει εφαρμόσει αυτά τα συμπεφωνημένα. Θέλει να ξαναγραφτούν οι κανόνες πριν μπει στη λέσχη. Αν έχουμε αρχές εδώ στο Κοινοβούλιο πρέπει να δώσουμε σαφές μήνυμα στην Ισλανδία. Η συμπεριφορά της για το γάδο είναι απαράδεκτη. Είναι απαράδεκτο προηγούμενο για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κατόπιν να αγνοήσει η Ισλανδία την πληθώρα άλλων κανόνων της Ένωσης. Ευχαριστώ. Ντότζ. Είναι η κυρία Μπασέσκου. Ευχαριστώ. Ψήφισα υπέρ τη έκθεση Πρέντα γιατί προβαίνει σε πολύ ισορροπημένη αξιολόγηση της κατάστασης των διαπραγματεύσεων διεύρυνσης ε, για την Ισλανδία. Και οι μεταξύ αυτές διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να είναι πρότυπο ενταξιακών διαπραγματεύσεων έχουμε μια ε, βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και ίσω και ενίσχυση της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και βελτίωση των διατλαντικών σχέσεων. Μια τέτοια διεύρυνση θα συμβάλλει και στην ανάπτυξη της ακτικής πολιτικής ε, σε περιφερειακό επίπεδο. Η διεύρυνση προς την Ισλανδία θα έχει θετικά αποτελέσματα παρατηρώντα και τις ε, υπόλοιπες υποψήφιες χώρες να επιταχύνουν τη διαδικασία. Σημαντικό επίσης είναι το θέμα της ε, ενημέρωσης ε, του κοινού γιατί υπάρχουν υπάρχει μεγάλη διάσταση απόψεως στην Ισλανδία σε ό,τι αφορά τις... Ε, την ενταξιακή προοπτική. Επίσης θα πρέπει να παρατηρήσουμε την Ισλανδία να άρει τους περιορισμούς για τους... της Ρουμανίας που θέλουν να εργαστούν στη χώρα αυτή. Ο κύριος Καμίνσκι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ ψήφισα υπέρ της έκθεσης γιατί Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διευρυθεί. Θα πρέπει να διευρυθεί προς όλες τις χώρες που ενστερνίζονται τις αξίες μας, που είναι δημοκρατικές χώρες, που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, που τηρούν και σέβονται τους όρους ε, της ελεύθερης οικονομίας. Και σίγουρα η Ισλανδία είναι μια τέτοια χώρα. Κατά τη γνώμη μου και για μας την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να μας διδάξει η κατάσταση στην Ισλανδία τα τελευταία χρόνια. Πολύ βαθιά, άνευ προηγουμένου, χρηματοπιστωτική κρίση, αλλά ταυτόχρονα και πολιτική κρίση. Και θα πρέπει να διδαχθούμε και από τον τρόπο με τον οποίο εξήλθε από την κρίση η Ισλανδία. Πολλοί λοιπόν είναι οι λόγοι που συνηγορούν υπέρ της διεύρυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς την Ισλανδία. Φυσικά Αναφέρεται ότι για να χορέψει κανείς τάγκο χρειάζονται δύο παρτενέρ και για να γίνει η Ισλανδία μέρο, κράτος μέρος Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η δηλωμένη προς αυτό βούληση των πολιτών της Ισλανδίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Καμίνσκι. Περνάμε τώρα στην τελευταία έκθεση, την έκθεση σχετικά με τη διεύρυνση για Βοσνία ριζεγοβινη Το λόγο του κύριος Κούκαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπερψήφισα το ψήφισμα για την Βοσνία Ζεγοβίνη. Ελπίζω να αποστείλει κάποια μηνύματα για να αναλογιστούν οι πολιτικοί στη χώρα αυτή και να προωθήσουν τις μεταρρυθμίσεις που επιγόντως χρειάζεται η χώρα. Επίσης, υπογραμμίζω ότι έχει πρωταρχική σημασία οι πολιτικοί στην Βόσνια Ετζεγοβίνη να βρουν το κουράγιο, την πολιτική βούληση να συνεργαστούν. Πρέπει να υπάρξει μια πολιτική, μια κουλτούρα πολιτικού συμβιβασμού και επικοδομητικού διαλόγου. Υπάρχουν μεγάλα θέματα, συνταγματική μεταρρύθμιση, δικαστική μεταρρύθμιση, άλλες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Δεν μπορούν να γίνουν όλα αυτά χωρίς κοινέ προσπάθειες. Η πρόοδος ε, στη χώρα και η διαδικασία ενοποίησής της είναι προς το όφελος, προς το συμφέρον της ασφάλειάς μας, της ε, σταθερότητας της περιοχής, αλλά είναι υπέρ και των Ευρωπαίων και των πολιτών της χώρας. Ευχαριστώ κύριε Κουκάνη. Η κυρία Έλληνα Μπασέσκου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπερψήφισα την έκθεση αυτή γιατί ε, η μακρά πολιτική ε, εμπλοκή έχει ε, δημιουργήσει αρνητικές επιπτώσεις στη Βοσνία Ριζεγοβίνη Ευελπιστώ ότι η νέα κυβέρνηση θα προχωρήσει σε πολιτικές μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε να αποκαταστήσει το κράτος δικαίου και τις σωστές οικονομικές πολιτικές. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι μια καλή ευκαιρία έτσι ώστε η Βοσνία Ριζεγοβίνη να προοδεύσει στη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο κατά αυτή την έννοια και θα πρέπει να βοηθήσει τη χώρα χωρίς όμως να πάρει θέσεις τέτοιες οι οποίες ε, να υποδαβλήσουν τα πάθη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ε, επίσης ευελπιστώ ότι η πολιτική στο Σαράγεβο θα είναι τέτοια έτσι ώστε να ε, γίνει καλύτερη η πολιτική απέναντι στους Ρωμά. και επίσης το θέμα των ορυχείων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είχα βάλει ερώτηση σχετικά με αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τάνοκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως και όλη μου η ομάδα, εγώ υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με τη διεύρυνση για την Ποσνία Ζεγοβίνη. Πιστεύουμε ότι σε αυτήν την χώρα ζωτική σημασία υπάρχουν ε, σημαντικά αιτήματα όσον αφορά κυρίω ε, την κεντρική κυβέρνηση ε, και επίση στοιχεία τα οποία θα πρέπει να σεβαστεί η κυβέρνηση του Σαράγεβο πριν προχωρήσουμε. Πιστεύουμε ότι η περιοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αυξηθεί. Η προσπάθεια καταπολέμηση διαφθορά θα πρέπει να είναι σημαντική, κυρίω δε η διάρθρωση ε, του συστήματος εκπαίδευσης ε, και του δικαστικού συστήματος ε, καθώς επίσης και η προστασία των ανηλίκων είναι θέματα πάρα πολύ σημαντικά. Επίσης θα πρέπει να καταπολεμηθεί αυτή η αύξηση της νέα μορφή τρομοκρατίας την οποία βλέπουμε στην χώρα. Στην έκθεση αναφέρεται αυτό ριζοσπαστικοποιώντας ένα τμήμα του πληθυσμού απέναντι σε ένα άλλο δεν αποτελεί λύση για την αποκατάσταση Κατάσταση ειρήνη στην Βοσνία Ερζεγοβίνη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τάνοκ. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Μπίλ. Ευχαριστώ. Η Βοσνία Ερζεγοβίνη είναι η χώρα που κατεξοχή δειροπάθησε από, από το μακροχρόνιο πόλεμο των Βαλκανίων. Ακόμη και σήμερα, πολύ, ε, σε τακτά χρονικά διαστήματα, σπαράζεται από εσωτερικέ ε, διαταραχέ. Εν μέρει εξαιτία και τη έξαρση του βαχαμπητικού εξτρεμισμού δεδομένης περίπλοκης δομής της εξουσίας, χαιρετίζουμε με αισιοδοξία το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης και παροτρύνουμε για πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας και του διαλόγου για τις δημοσιονομικές διαδικασίες και την εφαρμογή των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων. Επίσης και η δέσμευση της, των Βρυξελών με τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του ειδικού εκπροσώπου επιτρέπει την διαθέτηση των εκκρεμωτήτων προκειμένου να ενισχυθεί να επιταχυθεί η διαδικασία προσχώρηση τη Βοσνία. Φυσικά θα πρέπει να διευθυνθεί και το θέμα των υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου και, τις, και να εξαλειφθούν οι τρομοκρατικέ απειλέ. Ε, χαιρετίζουμε την εντατικοποίηση των προσπαθειών των κυβερνήσεων Βοσνία, Σερβία και Κροατία προκειμένου να διευθετηθούν οι εκκρεμότητε και να ενισχυθεί η, διαπεριφερειακή ασφάλεια. Για όλου αυτού του λόγου στάχθηκα υπέρ του ψηφίσματο. Σα ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριο Καμίνσκι. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, η Βοσνία και η είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Λέω ανεπιφύλακτα ότι η Βοσνία είναι η τύψη συνείδησης της σύγχρονης Ευρώπης. Σε αυτή τη δημοκρατία, την πρώην δημοκρατία, έλαβαν χώρα ε, τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα που έλαβαν χώρα στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ε, ε, ανήμπορα κοιτούσαμε και δεν βοηθήσαμε τη χώρα αυτή παρόλο που βλέπαμε τα αποτρόπια εγκλήματα που συνέβαιναν εκεί. Είδαμε ε, να χάνουν ε, τα παιδιά τους οι κάτοικοι της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Είδαμε τα φοβερά αυτά εγκλήματα. Σήμερα η Βοσνία Ερζεγοβίνη θέλει να προσχωρήσει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πληρώσει το ηθικό χρέος που έχει προς την χώρα αυτή. Δεν θα πρέπει να τα βλέπουμε όλα ε, ε, Θα δημιουργηθούν προβλήματα, αλλά η, η προσχώρηση της ε, Βοσνίας θα ε, ενισχύσει και τον πλούτο μας. Υπάρχουν, είναι πολύ πολυθρησκευτική αυτή η χώρα. Θα πρέπει να επιτρέψουμε τη Βοσνία Ερζεγοβίνη να βρει τη συνέχειά της και να βρει τη θέση που της αξίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Καπίνσκι. Ο τελευταίος Εύαλ Στέτλα. Υπάρχουν πολύ σωστά στοιχεία στην έκθεση αυτή. Αναφέρεται το θέμα του βαχαμπισμού, του βαχαμπισμού και του Ισλαμικού φανατισμού. Άρα υπάρχουν ε, κίνδυνοι. Αλλά παρόλα αυτά υπερψήφισα την έκθεση. Δεν είναι δυνατόν να αποφασίσουμε εμείς εκ το εξωτερικό ποια θα είναι η, η κρατική οργάνωση. Άκουσα διάφορους να τα λένε αυτά. Επαναλαμβάνω, απ' έξω δεν μπορούμε να διατάξουμε τι θα κάνουν. Ούτε μπορούμε να την κάνουμε ένα μόνιμο προτεκτοράτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Εδώ και 20 χρόνια η χώρα αυτή δεν είναι σε θέση να δημιουργήσει δομές δεν είναι σε θέση ούτε καν να οργανώσει τις υποθέσεις για το 2012. Δεν μπορούν ούτε καν να ονομάσουν υπεύθυνους διαφόρων υπηρεσιών. Και από ό,τι άκουσα, προτείνεται να, τις επόμενες γενιές να γίνει ένα ενίο κράτος. Είναι λάθος η ευρωπαϊκή πολιτική για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Η συνεδρίαση διακόπτεται μέχρι τις 3 η ώρα.